Σα ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γεωργίβα. Ολοκληρώνεται εδώ η εκθέταση του θέματο. Η ψηφοφορία θα γίνει σήμερα στι 12 το μεσημέρι. Επόμενο σημείο τη σήμερας ε, διάδεξη. Η έκθεση κυρίας Ρέγκνερ όσον αφορά την διασυνολική μεταφορά τη έδρα εταιριών. Τέσσερα λεπτά έχει το λόγο η συγκέντρια. Παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Επίτροπε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω του κοιόδε συζητητέ για την επικοδομητική συνεργασία μαζί μου ιδίω τον κύριο Ζένα και την κυρία Τάιν, αλλά επίση και τον κύριο Βουλό που προετοίμασε την ομοδότηση στην Επιτροπή Απασχόληση, η οποία αναφέρει πάρα πολύ σημαντικέ πτυχές όσον αφορά το σχέδιο μεταφορέ και την συμμετοχή των εργαζομένων και των εκπροσώπων του. Η πρόταση έκθεση υιοθετήθηκε ομόφωνα στην Επιτροπή μας και με μεγάλη πλειοψηφία στην Επιτροπή Απασχόλησης. Αυτό σημαίνει ότι η Κομισιόν θα πρέπει πια να δράσει νομοθετικά. Το θέμα της έδρας ε, είναι πολύ σημαντικό, καθώς επίσης το θέμα της συμμετοχής των εργαζομένων. Μία ε, εταιρεία η οποία μεταφέρεται από μία χώρα στην άλλη έχει ένα τεράστιο πρόβλημα, δηλαδή θα πρέπει να διακόψει την ε, παρουσία σε μια χώρα και μετά να μεταφέρει σε μια άλλη χώρα. Και αυτό μέσα στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς. Κοστίζει δηλαδή κάτι τέτοιο χρόνο, χρήμα και νεύρα. Και σχετίζεται και με κοινωνικά προβλήματα. Υπάρχει δηλαδή ένα κενό εδώ διακανονιστικό και το ξέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το έχει πει πλειστάξει στο παρελθόν στην ε, Κομισιόν, καλώντας την να νομοθετικά. Οι επιπτώσει για τι επιχειρήσει είναι ποιε. Οι επιχειρήσει εξαφανίζονται. Υπάρχει δηλαδή ένα ανταγωνισμό των ε, κάστοτε εθνικών νομοθεσιών για, ε, για την πρόσκληση των εταιριών αυτών, ε, των ανωνύμων εταιριών περιορισμένης ευθύνης αυτό δεν επιτρέπεται. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια οδηγία για τι ε, εταιρείε όσον αφορά την διασυνολική μεταφορά της έδρας τους. Γιατί κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνεται όχι ε, στυλ καουμπόι αλλά με τάξη. Ε, Αλλιώ χάνονται πολλά καθοδόν. Δεν επιτρέπεται δηλαδή οι επιχειρήσει να εξαφανίζονται για να φύγουν από τις υποχρεώσεις που έχουν σε μια χώρα. Λοιπόν, καταρχήν, όσον αφορά το θέμα της ε, συμμετοχής των εργαζομένων. Η συμμετοχή των ε, εργαζομένων οδηγεί σε μία αηφόρο επιτυχία των ε, επιχειρήσεων. Τα δικαιώματα των εργαζομένων θα πρέπει να είναι βάση του κεκτημένου, δηλαδή να σέβονται οι εταιρείε ε, το δικαίωμα διαβούλευση, ενημέρωσης και συναπόφασης των εργαζομένων. Αυτό σημαίνει ότι καλείται η Κομισιόν να γίνουν διαπραγματεύσεις ούτως ώστε να μπορέσουν να προστατευτούν τα ισχύοντα δικαιώματα ε, στην απόφαση και επίσης εφαρμογή των ε, βελτίστων πρακτικών. Τώρα το θέμα της έδρας. Καυτό. Ορισμένες χώρες επιτρέπουν την ε, διάκριση μεταξύ της διαχειριστικής έδρας και της κεφαλογικής έδρας. Δεν γίνεται αυτό παντού. Η έκθεση σημειώνει ότι εμείς δεν θέλουμε μία φοροδιαφυγή, δεν θέλουμε τη δημιουργία επιχειρήσεων ε, ταχυδρομικής θηρίδας. Αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε μια πρακτική λύση. Στην έκθεση βρίσκουμε μια σολομονική λύση, κύριε Επίτροπε. Παρακαλώ πέστε στον κύριο Μπαρνιέ που είναι αρμόδιος το θέμα αυτό να δράσει επιτέλους και να δράσει για το κεντρικό θέμα. Δηλαδή την μεταφορά αυτή της έδρας όλους τους ε, τομείς που αφορούν όλα τα κράτη-μέλη και μπορούν να βρουν όλα τα κράτη-μέλη σύμφωνα. Δηλαδή, η εσωτερική αγορά μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη, πράγμα που χρειαζόμαστε σήμερα περισσότερο από ποτέ. Μην διστάσετε λοιπόν να υποβάλλετε μια πρόταση και μην επαναλάβετε τα σφάλματα που έγιναμε με τι ευρωπαϊκέ ιδιωτικέ εταιρείε. Ευχαριστώ. Πρώτα ευχαριστώ κύριε Ρέγνερ. Περνάμε αμέσω στο ΚΑΣΟΔΙΑΗ. Η κυρία Τικάου έχει το λόγο. transfrontalier al companiilor reprezintă Ευχαριστώ. Ένα από τα βασικότερα ζητήματα της εσωτερικής αγοράς είναι η διασυνοριακή λειτουργία των επιχειρήσεων, άρθρα 49 και 54 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ένωση, όπου προβλέπονται η ελευθερία για την εγκατάσταση των επιχειρήσεων. Όμως ε, για τη μεταφορά των εδρών των εταιριών ε, ισχύουν διαφορετικές νομοθεσίες ανάλογα με το κράτος μέλος για το οποίο μιλάμε ως προς τις διοικητικές ε, δυσκολίες παρατηρούνται μεγάλες διαφορές και ως προς το κόστος που συνεπάγεται τη μεταφορά. Επίσης δημιουργείται νομική ανασφάλεια και θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει μία πρόταση, ένα σχέδιο νομοθετήματος για τη μεταφορά των εδρών των επιχειρήσεων στο ιστορικό της Ένωσης. θα έπρεπε να γίνεται η μεταφορά κατόπιν διαβουλεύσεως με τους ε, εργαζομένους. Επίσης, οι μονοαπευθυντικές ε, θηρίδες, όπως και στην οδηγία υπηρεσιών, είναι ένα εργαλείο που θα μπορούσε να βοηθήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Τσικάου. Η κυρία Πλατσικόβα Μπένοβα, τελευταία για διαδικασία Κατσουδιάη. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Εκτιμώ ιδιαίτερος ε, τη δουλειά της κυρίας Ρέγνερ. Η μεταφορά εταιρικών εδρών ε, απαιτεί σωστή νομοθεσία. Φυσικά χρειάζεται ελευθερία για να αναπτυχθεί το επιχειρηματικό πνεύμα. Όμως, εάν ε, η μεταφορά των εδρών γίνεται, ολοκληρώνεται μέρικος ε, ε, θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει αυτό για τα φορολογικά συστήματα των κρατών μελών. Το θέμα των γραμματοκιβωτίων βιτρινών για εικονικές εταιρείες είναι ένα γνωστό πρόβλημα στην Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να προστατεύονται οι τίμιες εισαγωγικά εταιρείες γιατί θέλουν να δρουν ε, σύνομα όταν μεταφέρουν τις έδρες τους. Επίσης η χρησιμοποίηση ενός συστήματος ελέγχου με τη συμμετοχή των εργαζομένων θα μπορούσε να βοηθήσει θα έπρεπε να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια οι εργαζόμενοι. Ευχαριστώ, συνάδελφε κυρία Φλωσίκοβα Μπένοβα. Η Επίτροπος κυρία Γεωργίευα έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί βουλευτέ, θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Ρέγνερ και την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για την έκθεση σχετικά με τη διασυνοριακή μεταβίβαση των εταιρικών ευρών. Ε, είναι ιδιαίτερα επίκαιρη η έκθεση, διότι το Φεβρουάριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δρομολογήσει η δημόσια διαβούλευση για το μέλλον του εταιρικού δικαίου στην Ένωση. Άρχισε η διαδικασία με μια διάσκεψη που έλαβε χώρα το Μάιο του 2011, πέρυσι δηλαδή, και ακαδημαϊκοί, δήμονες, ε, ε, άνθρωποι από ε, διάφορες περιοχές ήρθαν εδώ στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν αυτά τα θέματα. Επίσης υπάρχει ομάδα εμπειρογνωμόνων που προετοίμασε τη διάσκεψη από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκτοτε συνεχίσαμε την εξέταση του θέματος. Ε, και διευρύναμε τον κύκλο των πολιτών που μετέχουν σε εργασίες ε, ε, σκοπεύοντας να δρομολογήσουμε όπως σας είπα το Φεβρουάριο μια ευρεία διαβούλευση. Δεν θέλουμε να περιοριστούμε σε μια οδηγία για τις κατακεχωρημένες έδρες των εταιριών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να έχουμε ένα ευρύτερο πλαίσιο στη διαβούλευση. Θα έχουμε λεπτομερείς ερωτήσεις σχετικά με όσους πρέπει να ισχύουν ενδεχομένω για να εγκριθεί κάποια σχετική οδηγία καθώς και για τις πιθανές επιπτώσεις ε, αυτές. Οι απόψεις ε, που περιέχονται στην έκθεση θα αξιοποιηθούν ε, από αυτήν τη διαδικασία διαβούλευσης. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Δεν είναι η πρώτη φορά που το Κοινοβούλιο ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει πρόταση για διασυνοριακή μεταβίβαση εταιρικών εδρών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη συμμετάσχει σε ένα διάλογο για να διαπιστωθεί ανάγκη έγκρισης μιας τέτοιας οδηγίας. Θα πρέπει να προσφέρει πραγματικά πραγματική προσθεμένη αξία και για τι εταιρείε και για την εσωτερική αγορά και ξεκάθαρα αυτό ε, το θέμα συνεχίζει να απασχολεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν δύο ειδικά ζητήματα στον τομέα αυτό που απαιτούν προσεκτική εξέταση. Αναφέρομαι εδώ πέρα στη διάκριση ανάμεσα στην κατακεχωρημένη διοικητική έδρα της εταιρεία αφενός και στην συμμετοχή των εργαζομένων αφετέρου. Οι διαπραγματεύσεις για, για το καταστατικό των ιδιωτικών ευρωπαϊκών εταιριών κατέδειξαν πόσο δυσχερεί είναι οι διαπραγματεύσεις για επίτευξη συμβαστική ε, ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ευγνώμων για την έκθεση αυτή και συνεχίζει και εκείνη τι προσπάθειε τη ε, στον τομέα αυτό. Θέλουμε να συνεχίσουμε λοιπόν τον επικοδομητικό διάλογο με το Κοινοβούλιο για αυτό το σημαντικό θέμα τη εταιρική κινητικότητα εν γέννη και για την οδηγία για τη διασυνοριακή μεταφορά ε, των εταιρικών αδρών. Όλο ιδιαίτερα σα διαβεβαιώ ότι ο Επίτροπος Μπαρνιέ θα αναλάβει προσωπικά και θα ενημερωθεί για τη σημερινή συζήτηση ε, θα ολοκληρώσουμε, η πρόθεσή μας είναι να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία ε, κατά το τρέχον έτος, κατά το 2012. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Γεωργίευα. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση του θέματο. Η ψηφοφορία θα γίνει σήμερα στι 12 το μεσημέρι. Το επόμενο σημείο τη ημέρα τη είναι η έκθεση του κύριου Νόιζερ σχετικά με τα αξιοποίηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση